Bonjour euh, et bienvenue à... Καλημέρα. Καλώς ήρθατε όλοι. Ξεκινάμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σας προτείνω να προσθέσουμε ένα σημείο στην ημερήσια διάταξη για να μας παρουσιάσει η Κομισιόν μία ανεξάρτητη έκθεση με τίτλο «Ευρωπαϊκή Έκθεση για την Ανάπτυξη 2011-2012» και θα γίνει παρουσίαση σήμερα το απόγευμα μετά από το σημείο 5 που είναι οι ερωτήσεις προς την Κομισιόν. Έχετε κάτι για την ημερήσια διάταξη όπως τροποποιήθηκε εγκρίνεται τότε έγκριση των αποφάσεων και συστάσεων των συντονιστών της 19ης Ιουνίου του 2012. Έχετε όλα τα στοιχεία στο φάκελό σας και αν έχετε παρατηρήσεις θα πρέπει να τις ε, αναφέρετε στη γραμματεία πριν από το τέλος της συνεδρίασης, αλλιώς εγκρίνονται. Εγώ δεν έχω καμία ανακοίνωση και πάμε στο σημείο 4 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε μία διπλή δήλωση της ε, Επιτροπής και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για την κατάσταση στη Γουινέα Μπισάου. Όπως γνωρίζετε, στις 12 Απριλίου έγινε ένα στρατιωτικό πραξικόπημα στην Γουινέα Μπισάου, το οποίο καταδικάστηκε ευρέως από την ε, διεθνή κοινότητα και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εγκρίναμε ένα ψήφισμα στις 13 Ιουνίου σχετικά. Ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να έρθει στην Επιτροπή μας για να μας αναφέρει πώς έχει κατάσταση σήμερα στη χώρα και η Κομισιόν να μας εξηγήσει τις επιπτώσεις του πραξικοπήματος στην συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πρωτόκολλο αλίας το οποίο υπογράψαμε με τη Γουινέα Μπισάου και που θα έπρεπε να αρχίσει προσωρινά να εφαρμόζεται στα μέσα Ιουνίου πριν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. Η συνάδελφος Γκέζιν Μάισνερ είναι η συγγήτρια της νομοδότης Επιτροπής μας για το πρωτόκολλο Αλίας. Δίνω το λόγο στην... στον κύριο Φερνάντο Πόνς της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως είπε και η Πρόεδρος, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε στεναρά το πραξικόπημα της Γουνέας Μπισάου στις 12 Απριλίου και ζήτησε στη συνέχεια να αποκατασταθεί η συνταγματική τάξη που σημαίνει δημοκρατικές εκλογές και κυρίως ε, η εξαφάνιση των στρατιωτικών από, την πολιτική, από τον πολιτικό βίο της Γουινέας Μπισάου. Ζήτησε να υπάρξει μια βαθιά μεταρρύθμιση του τομέα της, ασφαλή, της ασφάλειας, η ατιμορρησία έπρεπε να τελειώνει, όπως επίσης ε, και το λάθρεμπόριο ναρκωτικών που αποτελεί μάστιγα για αυτή τη χώρα πολύ περισσότερο από τις άλλες, θα έπρεπε να σταματήσει το συντομότερο. Η Κάθριν Άστον ήδη πολλές φορές τόνισε όλα αυτά τα σημεία και επίσης ε, τόνισε και την υποστήριξή μας για την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης στην Γουινέα Μπισάου. Εμείς έχουμε απόλυτη συνείδηση για το πόσο σύνθετη είναι η κατάσταση. Θα θέλαμε να έχουμε μία δημοκρατική λύση και ενωτική. Εμείς θεωρούμε ότι η μεταβατική κυβέρνηση σήμερα δεν είναι ούτε ενωτική, ούτε προχωράει στην διαδικασία εκδημοκρατισμού. Πρέπει να δούμε πώς θα απομακρυνθούν οι, στρατιωτικές δυνα... στρατιωτικοί από την πολιτική ζωή και το πώς ε, θα <coughs> παίξουν το ρόλο που ο στρατός θα πρέπει να παίζει κανονικά σε μια δημοκρατική κοινωνία. Ο Εμεί λοιπόν ω Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένουμε ότι θα πρέπει να έχουμε μια ενωτική διαδικασία που θα πρέπει να δεσμεύει όλες τις, ε, να συνενώνει μάλλον όλες τις πολιτικές παρατάξεις και θα πρέπει να αποκλείονται από αυτήν τη διαδικασία στρατιωτική. Ενθαρρύναμε όλους τους εταίρους μας να εργαστούν, να σταθούν στην 2040 κάθετος 12 ψήφισμα του ΟΗΕ για την ενωτική διαδικασία με benchmarks για την επανάστα... Ε, ε, ε, αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης. Σταμάτημα καταπολέμηση της ατιμορρησίας και του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Ολοκληρώνοντας θέλω να σταθώ στο θέμα της συνεργασίας. Σίγουρα οι συνάδελφοι της Κομισιόν θα σας τα πούνε αυτά αναλυτικότερα. Όπως γνωρίζετε, η συνεργασία με την ε, Γουινέα Μπισάου είχε σταματήσει ήδη μετά το πραξικόπημα του 2010. Εκτός από τα σχέδια εκείνα, τα οποία έχουν ε, άμεση σχέση με την υποστήριξη του πληθυσμού. Ξέρετε ότι η Βουινέα Μπισάου είναι από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, είναι η πιο φτωχή χώρα της Αφρικής. Έχουμε δυσκολίες και με τις συμφωνίες αλίας, αλλά για αυτά τα θέματα και με την αδειά σας ε, θα αφήσω την Κομισιόν να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριο Ριντουάν Αμπτουλραχμάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σα. 12 Απριλίου ήταν το πιο πρόσφατο πραξικόπημα στη Γουινέα βισαού και Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, απέσυρε αρχές Μαΐου ε, τη λειτουργία του ε, εθνικού διατάκτη. Επίσης έχουν ε, διακοπεί διαδικασίες συνεργασίες και τεχνικής υποστήριξης προς τα Υπουργεία. Στον τομεακό διάλογο στους ε, που καλύπτονται από την αναπτυξιακή συνεργασία επίσης έχει ανασταλεί η διαδικασία αυτή. Σχεδόν όλα τα έργα έχουν διακοπεί. Συνεχίζεται όμως η άμεση υποστήριξη στον πληθυσμό ε, από έργα που χρηματοδοτούνται από θεματικές γραμμές του προϋπολογισμού. Το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρωπίνα Δικαιώματα και το Μέσο Αναπτυξιακής Συνεργασίας εξακολουθούν να λειτουργούν στην κοινωνία των πολιτών, την υγεία, την ανάπτυξη της υπαίθρου και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτόν τον καιρό 40 είναι τα έργα που συνεχίζονται και επίσης έχουμε έρθει σε επαφή με εκείνους που τα εκτελούν για να βεβαιωθούμε ότι δεν υποστηρίζουν κυβερνητικούς οργανισμούς. Στα πλαίσια ε, της απόφασης 2011-492 ε, του Συμβουλίου είναι επιλέξιμη για τους στόχους της χιλιετίας η Γκινέα Γουινέα Μπισάου και ε, αναπτύσσουμε ένα πρόγραμμα 5,5 εκατομμυρίων για πρόσβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ε, εγγύων γυναικών και ε, παιδιών μέχρι την ηλικία των 5 ετών σε διάφορες περιφέρειες της χώρας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπαχ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα σταθώ στην Διευτική Συμφωνία με την Γουινέα Μπισάου. Η σχέση που έχουμε με αυτή τη χώρα για τα θέματα αλληλείας είναι παλιές σχέσεις και καλές σχέσεις, παρά τις πολιτικές δυσκολίες. Εμείς καταφέραμε να υπογράψουμε μια νέα συμφωνία αλληλείας για το Ιανουάριο του 2012 και αυτή η συμφωνία, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, ήταν μια καλή συμφωνία κατά τη γνώμη μου ανταποκρινόταν στους στόχους της αηφορίας, της ενίσχυσης των ελέγχων, της καλύτερης αποτελεσματικότητας και της ε, τομεακής υποστήριξης. Η υποστήριξη της, κοινής, ε, της ε, Μικτής Επιστημονικής Επιτροπής, τα μέτρα για τη μείωση του ανοίγματο των, των δικτύων, επίσης για τα VMS, τα πλογικά συστήματα, ρήτρες σχετικά με, τις, ε, την οικονομική συνεργασία. Παρουσιάζω σύντομα αυτή τη συμφωνία. Δεν άρχισε ακόμη να ισχύει. Θα σας εξηγήσω πού βρισκόμαστε, αλλά αυτή η συμφωνία ήταν μια καλή συμφωνία και για τα οικονομικά γιατί από 7,7 εκατομμύρια ευρώ περάσαμε στα 2,9 εκατομμύρια, στα 9,2 συγγνώμη. Καλύτερη, ε, μια καλύτερη συμφωνία που ανταποκρίνεται και στην αξία του αλλιεύματος στην περιοχή. Τώρα τον Απρίλιο μάθαμε κι εμείς όπως όλοι το πραξικόπημα Πληροφορήσαμε σχετικά τα κράτη-μέλη, δηλαδή τις επαφές μας στα Υπουργεία Ελίας και στο Συμβούλιο. Επίσης είχαμε και στενή επαφή με τις υπηρεσίες εξωτερικές και εξωτερικής δράσης και τις άλλες υπηρεσίες της Κομισιόν και επιτόπου με την αντιπροσωπεία μας και ε, συμπεράναμε ότι τα πλοία μας θα διέτρεχαν κίνδυνο άμα ψάρευαν στις, ε, όχθες της, ε, στις ακτές μάλλον της ε, Γουινέας Μπισάου. Οπότε δώσαμε οδηγίες στους τόλους μας να εγκαταλείψουν τα ύδατα της Γουινέας Μπισάου και να μην ψαρεύουν. Είπαμε λοιπόν να αναστείλουμε το πρωτόκολλο, ήταν ένα ετήσιο πρωτόκολλο το οποίο θα έλυγε στις 15 Ιουνίου αλλά η προθεσμία αναστολής όντας μικρή, ε, όταν, όντας ε, αυτή που είναι, είπαμε να το αφήσουμε να ξεψυχήσει μόνο του αυτό το πρωτόκολλο, μέχρι τις 15 Ιουνίου δηλαδή. Τώρα έχουμε αυτό το νέο πρωτόκολλο του Φεβρουαρίου, τριετές πρωτόκολλο, Συμφωνήσαμε λοιπόν με την Προεδρία και με την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να το φέρουμε στο Συμβούλιο αυτό το κείμενο και να το παρουσιάσουμε εμπρόθεσμα. Δηλαδή, αν έχουμε μία εξομάλυνση της πολιτικής κατάστασης, να ξαναπάρουμε το κείμενο και να θέσουμε ενισχύ το πρωτόκολλο. Εμείς έχουμε λοιπόν ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία, να παρουσιάσουμε δηλαδή στο Συμβούλιο το κείμενο και είπε το Συμβούλιο να παγώσει την εξέταση αυτού του νέου πρωτοκόλλου, δηλαδή Προς στιγμή τα τρία κείμενα σχετικά με αυτό το νέο πρωτόκολλο βρίσκονται στο τραπέζι του Συμβουλίου. Έχει ξεκινήσει τυπικά η εξέταση, αλλά δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση. Εάν δεν έχουμε δηλαδή την έγκριση και τον, το πράσινο φως από τους συναδέλφους που είναι επιτόπου και από την ΟΕΣ. Τώρα, Ο αρχηγός της αντιπροσωπείας μας στη Γουινέα Μπισάου έχει κάνει τη σχετική κοινοποίηση στις αρχές λέγοντας ότι δεν ε, έχει, έχουν έχουμε καταλήξει απόφαση στο Συμβούλιο και ότι από τις 16 Ιουνίου δεν θα υπάρχει καμία αλλιευτική δράση της Ένωσης αυτές της Γουινέας Μπισάου και επιμείναμε στα κράτη-μέλη ότι τα ευρωπαϊκά πλοιάρια δεν θα έπρεπε να τύχουν καμία ιδιωτικής άδεια από τις αρχές. Και είπαμε ότι αυτή η απόφαση θα πρέπει να γίνει σεβαστή και δεν θα ανεχτούμε καμία χώρα να ζητήσει άδειε αλίευσης εκτός του πλαισίου της συμφωνίας. Τώρα, για τις πληρωμές ε, από το πρωτόκολλο 2007-2011 έχουμε ένα χρέος, σχετικά δηλαδή με την τομεακή ενίσχυση είχαμε καθυστερήσεις και διορθώσεις και ένα άλλο τμήμα το οποίο είχε μειωθεί λόγω ορισμένων ανεπαρκιών. Βρήκαμε λοιπόν μια συμφωνία με τη Γουινέα Μπισάου για να πληρώσουμε γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και αυτό το, αυτή πληρωμή πάγωσε περιμένοντας μια βελτίωση της πολιτικής κατάστασης. Ολοκληρώνω. Ελπίζω να ήμουν εκτενής ε, και για την συμφωνία, αλλά και για το πρωτόκολλο το οποίο έχει παγώσει στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μάισνερ επιθυμεί το λόγο. Μάλιστα. Να πάρω το λόγο, δεν έχω πρόβλημα. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Τώρα περίμενα να ακούσω, να ξεραρχίσω από την αρχή. Έλεγα ότι είναι δύσκολη η κατάσταση και το γνωρίζουμε διότι υπάρχει μια συμφωνία που δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ και αυτό το καιρό η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει και άμεσο εταίρο συνομιλητή για να μπορέσει να υπογράψει συμφωνία. Αυτό αφορά και την ε, καθήλυνα αρμόδια Επιτροπή Αλίας, αλλά και εμά που γνωμοδοτούμε. Και από πλευρά αναπτυξιακή πολιτική θα πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε και εμεί τι μπορούμε να κάνουμε ή τι μας μένει πλέον να κάνουμε. Γιατί η μεταβατική κυβέρνηση που δεν ε, είναι ε, προϊόν νόμιμη διαδικασία, δεν μπορεί να θεωρηθεί από εμά τέρος. Θα τα αφήσουμε αυτό να εκπνεύσει, θα αφήσουμε τα έργα να τρέχουν για να υποστηρίξουμε τον πληθυσμό. Μα είπε ε, η Υπηρεσία εξωτερική δράση ότι 40 έργα παραμένουν ε, σε λειτουργία, όχι την αλληλεία, αλλά πράγματα, δημοκρατισμό, γεωργία, υγεία κτλ. Αλλά και η αλληλεία είναι κάτι το οποίο μπορεί να ε, αποτελέσει και αποτελεί πηγή εσόδων στη Γουινέα. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, όχι μόνο από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση και Επιτροπή Αλία, τα ύδατα στα ανοιχτά της Αφρικής ε, μειώνονται ε, ως πηγή αλλιευμάτων για τα σκάφη της Ένωσης, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό ότι θα πάμε εμείς να ψάρεψουμε και αλλά τι θα γίνει με τη χώρα. Θα πρέπει να κοιτάξουμε ε, έναν κοινό τρόπο λειτουργίας. Προς το παρόν δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω διαδικαστικό. Κυρία Λέβιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, έχω μερικές ερωτήσεις. Νομίζω ότι άκουσα να λέγεται ότι κάθε συνεργασία με τη Γουινέα Μπισάου το 2010 είχε διακοπεί εκτός από την αναπτυξιακή βοήθεια και αυτού του είδους την υποστήριξη. Θα ήθελα να, ε, να ξέρω γιατί οι συμφωνίες οι αλλιευτικές περιλαμβάνονται στην ε, συνεργασία ε, που συνεχίστηκε μετά το 2010. Γιατί όχι άλλα είδη εμπορικών σχέσεων ή άλλες δραστηριότητες εξεπλάγει όταν άκουσα ότι ο βασικός λόγος διακοπής των αλλιευτικών δραστηριοτήτων στην, στα ύδατα της Γνέας Μπισάου για λόγους ασφάλειας για τα κοινοτικά πλοία ε, και όχι από, λόγω μιας πολιτικής οδηγίας ότι θα έπρεπε δηλαδή να σταματήσουν οι δραστηριότητες μετά το πραξικόπημα. Θα ήθελα μερικές διευκρινήσεις για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ξαναδίνω και τον λόγο σε ένα από τα άτομα της Κομισιόν για να απαντήσει στην ερώτηση της κυρίας Λέβιν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αν κατάλαβα καλά, ένα από τα ερωτήματα ήταν για την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η άλλη για την Επιτροπή. Θα απαντήσω για την ερώτηση για την Υπηρεσία και οι άλλοι συνάδελφοι θα απαντήσουν για την ερώτηση που τέθηκε στην Κομισιό. Αν συμφωνείτε βεβαίως. Νομίζω ότι η ερώτηση ήταν και ευχαριστώ γι' αυτό σχετικά με την αναστολή της συνεργασίας, τη διακοπή. Νομίζω ότι το είπα, αλλά θα ήθελα να διευκρινίσω. Η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν μέρη ανεστάλλει μετά το πραξικόπημα του 2010. Αναφέρθηκα στην συνεργασία και όχι στις σχέσεις με τη χώρα. Και βεβαίως η αλλιευτική συμφωνία έχει βεβαίως μια διάσταση συνεργασίας αναμφίβολα, αλλά είναι επίσης ε, και μια αλλιευτική συμφωνία, μια εμπορική συμφωνία και μέρος ε, των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν διεκόπη. Ήταν μια συνεργασία που εν μέρη διεκόπη και κυρίως διεκόπη και ανεστάλλει στα τμήματα που θα μπορούσαν ε, να ωφελήσουν την κυβέρνηση, αλλά δεν διεκόπη, όπως είναι, είναι συνήθως η περίπτωση, ε, σε αυτές τις ε, περιστάσεις όσον αφορά την βοήθεια ε, που απευθύνεται στους πληθυσμούς. Αναφέρεται λοιπόν αυτή η διακοπή στην συνεργασία και όχι στις γενικές σχέσεις με τη χώρα όπου εντάσσεται στις σχέσεις αυτές η αληφτική συμφωνία. Ελπίζω να απήντησα στην ερώτησή σας. Ναι, σας δίνω τον λόγο, ναι, θα προσπαθήσω να συμπληρώσω εστιαζόμενο στην Αλλιευτική Συμφωνία το 2010 οι σχέσεις με τη χώρα αυτή κατέστησαν πιο δύσκολες λόγω της πολιτικής κατάστασης και την εποχή εκείνη διακόψαμε την διαπραγματευτική διαδικασία για την ανανέωση της αλιευτικής Συμφωνίας κατόπιν οδηγίας ρητής της κυρίας Δαμανάκη της Επιτρόπου μας και μετά κατά τη διάρκεια του 2011 ε, θελήσαμε μια νέα συμφωνία όσον αφορά στη δεύτερη παρατηρήση σας κυρία Λέβιν δηλαδή τα κίνητρα που μας οδήγησαν να ζητήσουμε από το στόλο από το μήνα Απρίλιο να αποχωρήσουν από τα ύδατα της Γουινέας Μπισάου. Βεβαίως η πολιτική κατάσταση έπαιξε το ρόλο της. Ίσως να κατέδειξα το, το, την, το επιχείρημα της ασφάλειας που ισχύει, διότι έχουμε ευθύνη απέναντι στο στόλο μας, απέναντι στα πλοία που πάνε να ψαρέψουν σε εχθρικά ύδατα καμιά φορά. Αλλά υπήρχε και το πλαίσιο το πολιτικό. Το πρόβλημα που είχαμε είναι ότι στον, στο ίδιο το πρωτόκολλο δεν υπήρχε βάση νομική που να επιτρέπει την ταχύτατη διακοπή, την απαιτούμενα ταχύτατη διακοπή ε, και αναστολή ε, της συμφωνίας της αλλιευτικής, διότι χρειάζεται ένας μήνας προειδοποίηση και θα πρέπει να αιτιολογηθεί αυτό το αίτημα για να επιτευχθεί αυτή η αναστολή ε, και η διακοπή της αλλιευτικής συμφωνίας. Εφόσον βρισκόμασταν τον Απρίλιο, ένα μήνα πριν από ε, δύο μήνες πριν από την, ε, το τέλος, την εκπνοή ε, και χρειάζεται προειδοποίηση για την διακοπή, σκεφτήκαμε να υιοθετήσουμε μια πιο ήπια λύση ζητώντας ευγενικά αλλά στεναρά στα κράτη-μέλη να αποσύρουν τα πλοία τους, πράγμα που έγινε με άμεσο τρόπο. Δεν νομίζω ότι ζητάει κανείς άλλο το λόγο. Α, η κυρία Μέισνερ. Ναι. Στην ε, Αλία ε, αυτό ίσχυε και οριστικά στα νυχτά της Γουινέας ε, Μπισάου. Είπαμε ότι είναι μία από τις πιο φτωχές χώρες και εκτός από τη Γεωργία η Αλία ε, είναι ένα προϊόν, μια πηγή εισοδήματος. Ε, γιατί έχουν και κάποια υποδομή εκεί ε, επεξεργασίας ε, προϊόντων που τα εξάγουν και είναι πηγή εισοδήματος. Τώρα δεν ψαρεύει κανείς εκεί. Και τι γίνεται με τους αλληλείς της χώρας, της ίδιας, όχι τα δικά μας σκάφη. Γιατί δεν έχουν τα πλεονεκτήματα που θα επέρεαν από τη συμφωνία. Μπορούμε να τους υποστηρίξουμε, όχι με νέα έργα, προφανώς όχι, για την αλληλεία, αλλά από δική σας πλευράς ε, της Γενικής Διεύθυνσης ΜΑΡΕ ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί μια τέτοια πρόταση διαδικαστική. Ξαναδίνω το λόγο στην Κομισιόν γι' αυτό. Φυσικά δεν έχουμε κανένα ευρωπαϊκό πλοιάριο που ψαρεύει σήμερα στα ύδατα της Γουινέας Μπισάου. Τώρα η παράκτια αλληλεία της Γουινέας Μπισάου συνεχίζεται, πρόκειται για ένα στολίσκο πολύ περιορισμένο που καλύπτει τις ανάγκες ε, της, ε, των τόπιων ε, δεν είναι ένας στόλος ο οποίος ε, έχει να κάνει με συνεργασίες ε, και συμφωνίες, πόσο μάλλον με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κατρίν δεν έχει παρατηρήσεις, κάποιος άλλος όχι. Σας ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη φάση. Δεν έχουμε λάβει ερωτήσεις για την Κομισιόν. Πάμε στο 5α. Παρουσίαση από την Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Έκθεσης για την Ανάπτυξη 2011-2012. Η Κομισιόν παρουσίασε πρόσφατα την Ευρωπαϊκή Έκθεση 2011-2012 για την Ανάπτυξη που αποτελεί και την βασική υλοποίηση της πρωτοβουλίας ε, κινητοποιούμε την ευρωπαϊκή έρευνα υπέρ των αναπτυξιακών πολιτικών που ξεκίνησε το, το 2007 και που υποστηρίχθηκε από την Κομισιόν και 7 κράτη-μέλη. Αυτή η ανεξάρτητη έκθεση εξετάζει βασικά θέματα που συνδέονται με την ανάπτυξη και τις ευρωπαϊκές προπτικές. Δύο από τους ε, συντάκτες της έκθεσης, ο κύριος Ντεβέλντε και ο κύριος Μάκη, είναι παρόντες. Σας παρακαλώ λοιπόν να μας παρουσιάσετε την εργασία σας και να οργανωθείτε για το πώς θα γίνει η παρουσίαση. Καλώς, ευχαριστώ πολύ. Dirk Ντεβέλντε λέγομαι και ήμουν επικεφαλής του έργου για την Ευρωπαϊκή Έκθεση για την Ανάπτυξη του 2012. Η έκθεση αυτή είναι μια έκθεση ανεξάρτητη και είναι η τρίτη έκδοση αυτή. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επτα κράτη-μέλη. Και αυτή είναι η τρίτη με τίτλο «Αντιμετώπιση ε, της πάνη σπάνιτος ε, είναι ε, τρία ε, Ινστιτούτα που έχουν καταρτήσει αυτή τη μελέτη ανεξάρτητα, 15 συντάκτες και 20 με 25 τα έγγραφα στα οποία βασιστήκαμε από την καλύτερη ευρωπαϊκή και άλλη έρευνα. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε στις 16 Μαΐου με τον Επίτροπο Πίμπαλξ και έκτοτε συζητούμε την έκθεση αυτή σε διάφορες πρωτεύουσες και είχαμε συζητήσεις και στα πλαίσια των στόχων για την αηφόρο ανάπτυξη στο Ρίο συν 20 εκεί στη διάσκεψη. Επιτρέψτε μου να σας δώσω μια επισκόπωση και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο. Σε 15 λεπτά θα σας παρουσιάσουμε αυτή την έκθεση. Στη διαχείριση των φυσικών πόρων, η πρόσβαση στο νερό, στην ενέργεια και στη γη είναι κρίσιμη για τη μείωση της φτώχειας. Στις πιο φτωχές χώρες υπάρχει πρόβλημα. 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια. Ε, ένα δις επίσης δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό. και επίσης έχουν και πρόβλημα υποσυτισμού όταν δεν έχουν πρόσβαση στη γη. Ταυτόχρονα η παγκόσμια κοινότητα ε, πιέζει πολύ τη χρήση των φυσικών πόρων και στην έκθεση αναφέρουμε ότι στα επόμενα 20 χρόνια η ζήτηση για νερό, για τρόφιμα και τα θα αυξηθεί 40 με 50% απλούστατα γιατί αυξάνεται ο πληθυσμός και το εισόδημά του. Αυτό υπονομεύει τις αναπτυξιακές προοπτικές των πιο φτωχών κρατών και μάλιστα των πιο φτωχών ε, ομάδων του πληθυσμού στα εσωτερικά των ε, κρατών. Ορισμένες κοινότητες, ας πούμε, αν δεν έχουν πρόσβαση σε νερό, ο κόσμος μεταναστεύει, εσωτερική μετανάστευση, πηγαίνει στο επόμενο χωριό για να βρει νερό. Τι λέγει λοιπόν η έκθεση, ότι θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις πιέσεις που εφίστανται οι φυσικοί πόροι και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να το ε, αναγνωρίσουν και να έχουν μια συνολική προσέγγιση σε αυτό. Ένα ολοκληρωμένο τρόπο αντιμετώπισης. Ε, γιατί ε, ονομάζουμε αυτή την προσέγγιση well από τα αρχικά στα αγγλικά του νερού, της ενέργειας και της γης θα πρέπει να αναλάβουν δράση και ε, πολύ ο δημόσιος τομέας, ο ιδιωτικός και η διεθνή κοινότητα. Και βεβαίως εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Να δούμε λοιπόν πώς συνδέεται αυτό το πλέγμα ε, του νερού, της ενέργειας και της γης. Μπορούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσει σα. Αν θέλετε περισσότερε πληροφορίε, μπορεί να απευθυνθείτε γραπτά και σε εμά και με email. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό το πλέγμα και η διασύνδεση των τριών πόρων, όχι μόνο επειδή είναι άρρηκτα συνδεδεμένα αυτά τα πράγματα, ε, οι πόροι, αλλά είναι πιο περίπλοκη η κατάσταση. Αυξάνεται η αλληλεξάρτηση. Αν περνάει κανείς από την χαμηλής ε, ε, ένταση σε γεωργία, στην υψηλή ένταση σε γεωργία χρειάζεται και περισσότερο νερό και περισσότερη ενέργεια και περισσότερη γη. Ε, επίσης, φεύγουμε από ένα κόσμο που ε, είναι σχετικά σπάνιοι οι φυσικοί πόροι και πάμε σε ένα κόσμο που είναι ε, απόλυτα σπάνιοι οι ανύπαρκτοι οι φυσικοί πόροι και επίσης η τιμολόγησή τους δεν είναι η σωστή. Ε, θα πρέπει να δούμε και με ποιο τρόπο χρεώνονται ε, αυτοί οι φυσικοί πόροι και τι γίνεται με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, κατά πόσον οι τιμές ανταποκρίνονται ε, στην πραγματικότητα και είναι κατάλληλες. Αυτό το πλέγμα λοιπόν των τριών ε, φυσικών πόρων που αναφέρουμε έχουν να κάνουν με το εισόδημα στα κράτη, με τον τρόπο που διαχειρίζονται τα ίδια τα κράτη αυτό, ας πούμε. Τα βιοκαύσιμα είναι σημαντικό παράδειγμα. Στην αρχή ε, θεωρούνται τα βιοκαύσιμα ένας τρόπος αντιμετώπισης ε, της ε, εξάντλησης του άνθρακα. γιατί θέλαμε να μειώσουμε την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Αλλά η παραγωγή βιοκαυσίμων επηρεάζει και ασκεί πίεση σε άλλους τομείς όπως το νερό και τη γη το έδαφος. Ε, τι έμαθα εγώ διαβάζοντας αυτά τα παραδείγματα. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε τομεακά, κάθετα. Ε, χρειάζεται μια συνολική προσέγγιση. Και όχι να θέλουμε να μεγιστοποιούμε έναν τομέα, αλλά να βελτιστοποιούμε μια ολόκληρη σειρά, ένα φάσμα τομέων. Αυτό είναι και η προσέγγιση νέξου στο πλέγμα που αναφέρουμε έτσι στα αγγλικά. Οι προτάσεις, είπαμε, μάλλον που δέχονται φυσικοί πόροι, υπονομεύουν και την βιώσιμη και η φόρο ανάπτυξη. Θα πρέπει η παγκόσμια κοινότητα να απαντήσει σε αυτό και στους εξής τέσσερις πυλώνες. Πρώτον, να διαχειριστούμε τη ζήτηση ε, φυσικών πόρων. Στο παρελθόν τι είδαμε. Όταν αυξανόταν το εισόδημα, το παγκόσμιο, αυξανόταν και η ζήτηση φυσικών πόρων. Ε, με λιγότερους ρυθμούς, χαμηλότερους, αλλά αυξανόταν. Και αν αυτό το προβάλλουμε στο μέλλον, κάποια στιγμή θα εξαντληθούν οι φυσικοί πόροι. Ε, θα πρέπει να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου να αυξάνεται με το εισόδημα και των φτωχοτέρων, αλλά να περιορίζεται όσο γίνεται η ζήτηση ε, φυσικών πόρων. Να χρησιμοποιούμε με φιδό αυτούς τους πόρους. Άλλο που πρέπει ε, να σκεφτούμε είναι η αύξηση της προσφοράς προς τους πιο φτωχούς. Ε, ενέργεια ανανεώσιμη, ενέργεια, ε, αποθήκευση νερού και πρόσβαση στη γη. Τρίτον, πώς θα βγούμε από αυτές τις προκλήσεις. Με καινοτομία, με αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων. Και ο τέταρτος πυλώνας είναι να βεβαιωθούμε ότι κάποιες χώρες και μάλιστα πιο φτωχοί στις χώρες ε, θα πρέπει να έχουν αντιστάσεις στις ε, διάφορους ε, κραδασμούς και κλειδονισμούς που ξαφνικά αντιμετωπίζουν. Έρχομαι τώρα στην επόμενη διαφάνεια που είναι μια σύνοψη του φάσματος δράσεων που προτείνουμε και που θεωρούμε σημαντικές για να αντιμετωπίσουμε τους ε, πόρους που σπανίζουν. Σας είπα, ζήτηση, προσβορά, ε, αποτελεσματικότητα και αντίσταση. Και τι δράσεις τώρα μπορούν να αναλάβουν διάφοροι φορείς. Ο δημόσιος τομέας, οι κυβερνήσεις δηλαδή, βεβαίως παίζουν εδώ σημαντικό ρόλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται μια χώρα Σκεφτείτε ε, πόση πίεση δέχεται, ας πούμε, η γη γιατί χρειαζόμαστε ε, μέχρι το 2030 ή το 2050 να ταΐσουμε ένα πληθυσμό που θα έχει ξεπεράσει τα 9 δισεκατομμύρια επίσης και για λόγους αεφορίας και βιοπικιλότητας και χρειάζεται και περισσότερη γη για ε, την καλλιέργεια φυτών για παραγωγή βιοκαυσίμων. Αυτές τις πιέσεις λοιπόν για τη χρήση γης θα πρέπει πρώτα απ' όλα να τις διαχειρίζονται τα κράτη. Άρα ο δημόσιος τομέας παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, ε, συντονιστικό κυρίως και ρυθμιστικό, ε, θέτοντα το σωστό ρυθμιστικό πλαίσιο. Ο ιδιωτικός τομέας παίζει σημαντικό ρόλο γιατί έχει ε, και περισσότερες δυνατότητες. Ε, με τρόπους φιλικούς προς το περιβάλλον είναι ευκαιρία αυτή για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και παντού ε, μπορούν να συνεργάζονται αυτοί οι φορείς σε ένα φάσμα δράσεων και δραστηριοτήτων. Ένα μόνο ανέφερε εδώ να αυξηθεί η πρόσβαση στην ενέργεια που είναι μεγάλη και σημαντική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ας πούμε για, στην ατζέντα για ε, αλλαγή και μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνδυάσει τα διάφορα μέσα που έχει, την τεχνική υποστήριξη της γνώσης που διαθέτει και να το συνδέσει με έναν τρόπο για να δημιουργηθούν εταιρικές σχέσεις και συνεργασίες με τις αναπτυσσόμενες χώρες για πρόσβαση στις ανανεώσιμες. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Τζέιμς για να σας εξηγήσει τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζοντας από την τελευταία διαφάνεια, τη μεσαία στήλη που έχουμε εδώ, που δείχνει σαφώς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ρόλο να παίξει σε πολλούς από αυτούς τους τομείς. Όλοι αυτοί οι τομείς έχουν μια κοινοτική διάσταση. Και τώρα εδώ σε αυτήν την διαφάνεια προσπαθούμε να διευκρινίσουμε, να προσδιορίσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορους τομείς. Πρώτα απ' όλα πρόκειται για την συνεκτική πολιτική με την ανάπτυξη. Υπάρχει μια κατηγορία εσωτερική πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να εξεταστεί. Έχουμε εδώ τα παραδείγματα που περιλαμβάνουν θέματα κατανάλωσης, αποδοτικότητα που έχετε ήδη στην Ευρώπη, ε, ένα θέμα επίμαχο και επίσης επίκαιρα θέματα όπως ε, η κοινή αγροτική πολιτική αναθεώρησή της και τα παραδείγματα βιοκαυσίμων που σας έδωσε ο προλαλής σας στις εξωτερικές πολιτικές που έχουν, που έχουν ε, επιπτώσεις προς τα έξω, που είναι το εμπόριο και οι επενδυτικές πολιτικές. Μπορείτε να βρείτε και άλλους τομείς, αλλά αυτοί είναι οι δύο βασικοί τομείς που ενέχουν σημασία κατά τη γνώμη μας, κυρίως επενδυτική πολιτική ε, σε τομείς ε, όπως είναι οι νέες υποδομές, καινοτομία κλπ. Και επίσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μετά υπάρχει μια κατηγορία συνεργασίας αναπτυξιακής Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ εξετάσαμε αναφορές ε, στην ατζέντα για αλλαγή, ε, στην ε, εταιρικέ σχέσεις για ανάπτυξη, που δείχνουν πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τους διάφορους τομείς που είναι σημαντικοί Ε, για το θέμα και στην επόμενη διαφάνεια έχετε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά υπάρχει ε, και το θέμα της διαμόρφωσης της παγκόσμιας ε, διακυβέρνησης και θα έχουμε μια συζήτηση για το Ρίο ΣΥΝ 20 για την Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον, θέματα που ξεπερνούν τα εθνικά σύνερα, τα υπερβαίνουν, που παίζουν σημαντικό ρόλο στον τομέα αυτών. Αυτό που έχετε εδώ είναι ένας κατάλογος τομέων στην αναπτυξιακή συνεργασία που μπορείτε να εξετάσετε. Δεν πρόκειται να διαβάσω όλους αυτούς τους τομείς, συνοψίζονται ε, στην ε, σύνοψη που έχετε σε ένα έγγραφο που βρίσκεται στην είσοδο της αίθουσας αυτή. Τα δύο τελευταία θέματα έχουν σχέση ε, με την διακυβέρνηση, την ολοκληρωμένη προσέγγιση, την διαφάνεια, τέτοια θέματα είναι ένα πακέτο βελτίωση της διακυβέρνησης στις αναπτυσσόμενες χώρες και πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια με συνεργασία, με εταιρική σχέση που είναι ε, σημαντική, ορισμένα σημεία σημαντική εταιρική σχέση διαμέσου των κυβερνήσεων και στον ιδιωτικό τομέα όπου υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, πολλές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα ε, συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο τη σημασία αυτών των θεμάτων και προσπαθούν να τα προωθήσουν εταιρικές σχέσεις και με άλλες οργανώσεις, με οργανώσεις πολιτών κλπ. Δεν έχουμε διερευνήσει όλες τις δυνατότητες, αλλά νομίζουμε ότι έχει σημασία η εταιρική σχέση με τον ιδιωτικό τομέα και υπάρχουν και ορισμένοι τομείς πολιτική σημαντικοί όπως είναι η περιφερειακή ολοκλήρωση, επίσης απαιτήσει πολιτικής ε, για θέματα διασυνοριακά που δεν σχετίζονται μόνο με μια χώρα, δεν είναι ε, δυνατό να τα αντιμετωπίσει κανείς με τον τρόπο αυτό, ε, με, ας παίρνουμε χάρη διαχείριση ύδατος σε μια λεκάνη απορροής, είναι ένα θέμα περιφερειακής ολοκλήρωσης, περιφερειακής προσέγγισης και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε θέση να μπορέσει να αντιμετωπίσει τέτοια προγράμματα ολοκλήρωσης και ένταξης περιφερειακής για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη το θέμα της μείωσης της φτώχειας. Βεβαίως, ίσως το θέμα αυτό να θεωρείται περιβαλλοντικό, αλλά είναι θέμα ατζέντα της φτώχεια, διότι οι φτωχοί είναι οι άποροι είναι αυτοί οι οποίοι επηρεάζονται πιο πολύ από την έλλειψη ύδατος κλπ. Το θέμα λοιπόν της μείωσης της πτώχειας, αυτή η διάσταση είναι εξαιρετικά σημαντική και τέλος όταν προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τα, τους τομείς κλειδιά, τα πολιτικά μηνύματα, τα βλέπετε είναι πέντε προτεραιότητες για δράση στον πολιτικό τομέα που είναι οι πιο σημαντικές και βλέπετε ότι η πρώτη έχει σχέση με την κατανάλωση. Μήνυμα για την Ευρώπη να εξετάσει αυτό το επίμαχο και δύσκολο θέμα, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να βελτιωθεί από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά. Επίσης, αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην καινοτομία σε πάρα πολλούς τομείς, παραγωγικότητα, γεωργική και αυτό δεν σημαίνει ε, μόνο υψηλή τεχνολογίας ε, γεωργία, αλλά επίσης ε, και με χαμηλή τεχνολογία. Δεν επιλέγουμε ένα σύστημα γεωργία σε σχέση με τα άλλα, την εντατική γεωργία. Ε, ίσως ή της χαμηλής ε, έντασης ε, την οικογενειακή γεωργία. Επίσης η παραγωγή ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντική. Να ασχοληθούμε με τους σπόρους αυτούς που σπανίζουν και πάλι στο τρίτο σημείο επανερχόμαστε στους θεσμούς, στους κανόνες του παιχνιδιού με το πώς κανείς προσεγγίζει το θέμα, την ικανότητα διαχείρισης των πόρων αυτών με τρόπο ολοκληρωμένο Πολλές οργανώσεις έχουν δημιουργηθεί από διάφορα υπουργεία και ε, υπηρεσίες για διάφορους τομείς, αλλά χρειάζεται μια συνολική προσέγγιση. Επίσης, αυτό που είναι ε, σημαντικό είναι η προώθηση πολιτικής της γης που να περιλαμβάνει όλους, να μην αποκλείει κανέναν, να μπορούν όλοι ε, να υψώσουν τη φωνή τους, να εισακουστούν ε, και συστήματα γης ε, τα οποία να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πιο ευάλωτων. Επίσης το θέμα της τιμολόγησης των φυσικών πόρων και των υπηρεσιών ε, με τρόπο περιεκτικό, συνολικό και θα δώσω και πάλι τον λόγο στον προλαλήσαντα για τα, τις τελικά συμπεράσματα και φθάνω στο τελευταίο αυτό σημείο της τιμολόγησης των φυσικών πόρων και υπηρεσιών που είναι ένα θέμα θεμελιώδους σημασίας και έχουν ξοδευτεί ένα 3 εκατομμύρια δολάρια σχετικά με τις επιχορηγήσεις αυτές για το περιβάλλον και στην Ευρώπη έχουν εξοδευτεί πάρα πολλά κονδύλια τα οποία εντείνουν τον τρόπο με τον οποίο ασχολούμεθα με την γεωργία ε, με έμφαση στο περιβάλλον. Όταν ε, εκπονήσαμε την έκθεση είχαμε και ένα βίντεο με ένα παράδειγμα για ε, το πώς ασχολούμεθα με το περιβαλλοντικό κεφάλαιο ας σκεφτούμε ε, πώς μπορούμε να κάνουμε πράγματα σε μικρότερη ε, κλίμακα. Έχουμε την Λιμνή στην ε, Κένια, όπου στα κατάντι οι χρήστες μπορούν να αντισταθμίσουν, να αποζημιώσουν κατά κάποιο τρόπο αυτούς που βρίσκονται στα ανάντι. Ελπίζουμε ότι το έγγραφο αυτό είναι ζωντανό με την έννοια ότι είναι σημαντικό για την ε, τεκμηρίωση της αλλαγής, ε, για τις αλλαγές που θα επέλθουν ε, και επίσης σημαντικό στα πλαίσια του Ρίο Συνήκωση και την παρακολούθηση για την διατύπωση της εξωτερικής ανάπτυξης, πολιτικής εξωτερικής ανάπτυξης. Είχαμε διάφορα άτομα, διαπραγματευτές, άτομα της Κομισιό και από την Παγκόσμια Τράπεζα και όλοι ε, συμφωνήσαμε ότι το είδωρο, η ενέργεια, η γη, τα τρόφιμα είναι πάρα πολύ ε, σημαντικά για τους στόχους μας και ε, θέτουμε στόχους που δεν είναι μόνο περιβαλλοντικοί. Σκεφτόμαστε όχι μόνο τη ζήτηση αλλά και την προσφορά και την κοινωνική πτυχή των στόχων και την αποδοτικότητα επίσης, τα οικονομικά δηλαδή του πράγματος και την ε, περιβαλλοντική πτυχή. Ελπίζουμε λοιπόν ε, ότι το έγγραφο αυτό είναι ζωντανό και περιμένω τις ερωτήσεις που έχετε να μας ε, θέσετε και ίσως και τα στελέχη της Κομισιό έχουν να προσθέσουν κάτι ως προς το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Κύριε Γκάραντς, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Έχω δύο ερωτήσεις προς τους ομιλητές. Η πρώτη αφορά στην πρόσβαση στη γη στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και αναφέρω εδώ δύο χώρες οι οποίες είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες γι' αυτό. Την Ζιμάμπουε και την Αμίμπια. Στην ε, Ζιμάμπουε Είδαμε τα αποτελέσματα μιας κυβερνητικής πολιτικής που απογυμνώνει τους ιδιοκτήτες, ε, τους γεωκτήμονες από τη γη τους. Αποτέλεσμα δεν υπάρχει παραγωγή και οι φτωχοί δεν έχουν τίποτα να φάνε. Η αντίδραση λοιπόν δεν ήταν καλή. καλή. με τα γνωστά αποτελέσματα. Στην Ναμίμπια είχαμε μία αντίστοιχη προβληματική, αλλά δεν ε, είχαμε τα ίδια επακόλουθα. Τι, πώς, μπορούμε εμείς ε, να αντιμε... πώς μπορούμε εμείς αντιμετωπίσουμε την κατάσταση όταν έχουμε μία αγροτική επανάσταση. Μήπως θα έπρεπε εμείς ε, να διαπραγματευτούμε με αυτές τις χώρες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αγοράσουμε τη γη από τους γεωκτήμονες. Βέβαια πρέπει να δούμε ποιος θα την πληρώσει αυτή τη γη. Να μην αφήσουμε δηλαδή να εξελιχθεί αυτό σε σύγκρουση. Και τελευταίο, είπατε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ΚΑΠΑ γίνεται όλο ένα και πιο σημαντική. Μα τι σας κάνει εσάς να λέτε τέτοιο πράγμα όταν ας πούμε τα κράτη ε, μειώνουν την παραγωγή και λόγω της μείωσης δηλαδή της χρήσης των νητρικών αλλά και σε εθνικό επίπεδο ε, μειώνουν την παραγωγή για να αποφύγουν τη χημική μόλυνση. Τέλος πάντων, για να, τα πω, για το πω αλλιώς, ότι όλες οι μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ τα τελευταία χρόνια ε, ήταν ε, ε, μεταρρυθμίσεις οι οποίες ε, δεν είχαν να κάνουν με τις εντατικές παραγωγές. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι, λέει η Πρόεδρος. Στα πλαίσια της μελέτης σας, υπολογίσατε τα απαραίτητα εκτάρια που χρειάζονται για να ανταποκριθούμε στις ανά, ενεργειακές ανάγκες, δηλαδή όταν μιλάμε εμείς για το biofuel, το έχετε, έχετε μετρήσει όταν μιλάτε για εντατικοποίηση της γεωργίας, έχετε υπολογίσει τους ιδρικούς πόρους που χρειάζονται για αυτού του τύπου τη γεωργία. Τώρα για την ε, ίδρυψη βλέπετε ότι έχουμε ένα σωρό φράγματα που χτίζονται στην, στην Αμαζονία για παράδειγμα με το θέμα της ε, εξάτμισης μήπως θα έπρεπε να αναθεωρήσουμε την πολιτική των, για την οικοδόμηση των φραγμάτων, ας πούμε δείτε το φράγμα του Ασουάν, όπου η εξάτμιση απορροφά το 40% του νερού. Μήπως πρέπει να το ξαναξαναδούμε αυτή την πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο η κυρία Σαρλότ Μπιουέ. Δεν είναι εδώ. Εδώ, εδώ είμαι. Φρανσουάζ Μωρό με λένε. γιατί η διαδικασία της Ευρωπαϊκής Έκθεσης ξεκίνησε πριν απο τρια τρία-τέσσερα χρόνια και ο στόχος ήταν να ακουστεί καλύτερα η φωνή των Ευρωπαίων ερευνητών στο διεθνές προσκήνιο ξεκινώντα δηλαδή από τη λογική ότι δεν υπάρχει ένα μονοπόλιο σκέψη για τι ανεπτυξιακέ πολιτικέ στη Ουάσιγκτον ή στη Νέα Υόρκη ή αλλού. Και δεύτερο στόχο είναι να έχουμε αυτόν τον τακτικό διάλογο και αυτές τις τακτικές ανταλλαγές με τα ευρωπαϊκά κέντρα, ε, ερευνητικά κέντρα, τα οποία έχουν τεράστιο δυναμικό, αλλά εργάζονται συνήθως μέσα από μια οπτική διάσταση και θελήσαμε να τους δώσουμε μια ευρωπαϊκή διάσταση για τις αναπτυξιακές πολιτικές. Αυτή είναι η τρίτη έκθεση ε, για την, ε, για διαχείριση των φυσικών πόρων και είναι ιδιαίτερα εύστοχη στην σημερινή διαδικασία με τις, προοπτικές, με τις πολιτικές προτεραιότητες που έχουμε, με τις πολιτικές για το περιβάλλον, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τον επόμενο κύκλο προγραμματισμού, για τη γεωργία, εμείς δεν έχουμε επενδύσει επαρκώς τα τελευταία χρόνια στο γεωργικό τομέα και όπως γνωρίζετε αυτή είναι και μία από τις προτεραιότητες μας για το μέλλον. Αυτή η έκθεση μας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και εύστοχη σήμερα. Επίσης είναι πάρα πολύ χρήσιμη και για τις ε, πολύ χρήσιμη αυτή η συζήτηση και για τις επόμενες ε, προοπτικές ε, για τις ΟΜΔ και για τη μείωση της στόχιας. Και να βρούμε οργανισμό Και να βρούμε λοιπόν ε, την, την κοινωνική διάσταση της αηφόρου ανάπτυξης. Ξαναδίνω το λόγο στους εξπέρ, στους εμπειρογνώμων. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πολύ σημαντικές ερωτήσεις και συγκεκριμένες. Αναφερθήκατε σε διάφορα σημεία να αρχίσω πρώτα. Η πρόσβαση στη γη είναι σημαντικό και τονίζουμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία όντω η διακυβέρνηση. Αλλά όταν δεν είναι σωστή αυτή, τι γίνεται. Ε, μιλάμε για πολλά τέτοια θέματα στην έκθεση και στα παραστήματα και είναι πολύ σημαντικό ε, να διαπιστώσουμε ότι οι χώρες που διαχειρίζονται σωστά τους φυσικούς τους πόρους το κάνουν όταν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν την ηγεσία αλλά και και ε, σωστές ε, πολιτικές αποφάσεις όταν λαμβάνονται. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε έξωθεν ε, κάπως συντονιστικά ή να επισημαίνουμε διάφορα στοιχεία της έρευνας ε, να κάνουμε κάποια μητρώα ε, συναλλαγών που έχουν να κάνουν με αγοραπολισία γης και κάποιες ε, κατευθυντήριες γραμμές εθελοντικές, ας πούμε, του ΦΑΟ για το πώς γίνονται οι αγοραπολισίες γης. Είναι σημαντικό αυτό γιατί αυξάνονται συνεχώς οι πιέσεις για τη γη και η ζήτηση και στο μέλλον θα αυξηθεί και η σημασία της γης. Εκεί είναι πολύ σημαντικό να το ξανασκεφτούμε και να προβληματιστούμε. Έγινε και μια ερώτηση για τα βιοκαύσιμα. Δεν έχω τα ακριβή αριθμητικά στοιχεία αυτή τη στιγμή στα χέρια μου. Στην έκθεση ε, έχουμε ένα πίνακα που αναφέρει όλα αυτά τα στοιχεία και θα βεβαιωθώ ότι θα τα λάβετε. Αλλά αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι σε ορισμένες χώρες η παραγωγή βιοκαυσίμων έρχεται ακριβώς σε ανταγωνισμό με άλλες χρήσεις της γης και αυξάνει και, την τιμή της γης. Σε άλλες χώρες δεν συμβαίνει αυτό απαραίτητος Να δούμε και ποιες είναι οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των βιοκαυσίμων ή και τι ε, πόρους και τι σχέσεις έχουν οι χώρες. η Βραζιλία έχει πολύ γη και πολύ νερό, ενώ η Κένια ε, για να συμφέρει η καλλιέργεια φυτών για παραγωγή βιοκαυσίμων θα πρέπει ε, να μην είναι εις βάρος της παραγωγής τροφίμων. Δηλαδή είναι ανταγωνιστικές αυτές οι καλλιέργειες μεταξύ τους. Γι' αυτό σας είπα ότι χρειάζεται μια ε, συνολική προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη αυτό το πλέγμα και των σχέσεων που έχουν ε, μεταξύ τους ε, το νερό, η γη και η ενέργεια. Έγινε ένα σχόλιο για την κοινή γεωργική πολιτική. Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή η έκθεση είναι αναπτυξιακή. Δεν είναι αναγκαστικά ιδιαίτερη έμφαση στην κοινή γεωργική πολιτική. Εκεί γίνεται έρευνα αλλού σε άλλο πλαίσιο που μπορείτε να αντλήσετε τα συμπεράσματα. Η έκθεση αυτή δεν αφορά την κοινή γεωργική πολιτική. Απλώς ήθελα να πω ότι θα πρέπει και αυτό να το δούμε σε ένα συνολικό πλαίσιο και τον τρόπο με τον οποίο επιδοτούμε ε, κάποιες δραστηριότητες, κάποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες, ας πούμε και τη χρήση των φυσικών πόρων. Και υπάρχουν τέτοια προγράμματα που προάγουν την ε, εκτατικοποίηση είναι ε, ευπρόσδεκτα, αλλά θα πρέπει να αλλάξει η όλη γεωργία από την εντατική να περάσει στην εκτατική. Δεν είμαι βέβαιος ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει πάντα. Προς το παρόν. James. Ναι, βεβαίως. Σχετικά με το σημείο του κ. Γκόραντς, ε, σχετικά με την πρόσβαση στη γη Νομίζω ότι η περίπτωση της Ζιμπάμπουε είναι μοναδική και αρκετά έντονη. Αυτό που είδαμε εκεί ήταν ακριβώς μια περίπτωση η οποία δεν είναι τελείως διαφανής και ένα από τα επιχειρήματα που προτάσσονται είναι ότι θα έπρεπε να καταστεί δυνατόν για την κυβέρνηση και τις δημόσιες αρχές να έχουν ε, διαδικασίες για τη γη, για τη μεταβίβαση γης, ε, η ε, διανομή γης που να επιτρέπουν προσφυγή στη δικαιοσύνη, που να επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μπορεί κανείς να εξετάζει την περίπτωση της Ζιμπάμπουε. Νομίζω ότι αυτό που θέλουμε να τονίσουμε εδώ είναι το θέμα της πρόσβασης με διαφάνεια. Όπως αναφέρθηκε, υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές της ΦΑΟ και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004 ήδη, που ε, αναδεικνύουν και τονίζουν ε, τη σημασία αυτών των χαρακτηριστικών. Ένας από τους λόγους για τους οποίους ε, εξετάσαμε έτσι το θέμα της γης ήταν ήταν η συνολική γενική ε, τάση, αυτή η τάση αύξησης αγορών ε, γης στην Αφρική κυρίως, που οδήγησε ε, σε μία μια, στη Μαδαγασκάρη όπου έχουμε την πολιτική διαδικασία που κάπως επηρεάζεται και έχουμε Υπάρχουν ε, άτομα σε διάφορα στη γη που, ε, των οποίων η γη πουλιέται χωρίς να έχουν καμία γνώση ότι πουλήθηκε η γη τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ζήτηση που αυξάνεται διεθνώς για τη γη. Δύο, ο τρόπος όπου αντιμετωπίζεται το θέμα αυτό πρέπει να είναι πιο διαφανής και πιο προσεκτικός ε, και θα πρέπει να βλέπουμε το θέμα όχι μόνο από την άποψη της γης αλλά και από την άποψη του ύδατος που υπάρχει εκεί. Αυτά είναι τα θέματα σχετικά με τη γη και την πρόσβαση στη γη. Για το θέμα των φραγμάτων. Ναι, τα φράγματα είναι ένας από τους τομείς όπου αυτή η διασύνδεση ανάμεσα στα τρία αυτά στοιχεία του WELL έχει σημασία, διότι το είδωρ ε, χρησιμοποιείται για την γεωργία, για την υδροηλεκτρική ενέργεια που είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας ε, και υπάρχουν και άλλα αιτήματα τα οποία είναι νόμιμα και αυτό που αναφέρατε ε, κυρία Πρόεδρε για την εξάτμιση του ύδατος που είναι και άλλο ένα θέμα. Ε, το είδωρ είναι πολύτιμο αν εξατμίζεται τότε αυτό με ορισμένα φράγματα, με φράγματα σε ορισμένα πλαίσια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να εξετάζεται. Αυτό για μας αντιπροσωπεύει ε, την ανάγκη ε, μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης. Δεν πρέπει κανείς να εστιάζεται μόνο στην ενέργεια ή στην ε, άρδευση. Θα πρέπει να εξετάζει κανείς τα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο. Αυτό βεβαίως δεν είναι μια απαγόρευση για την κατασκευή φραγμάτων αλλά πρέπει ε, να εξετάζεται κάθε κατάσταση ε, ως ιδιαίτερη κατάσταση μέσα στο δικό της πλαίσιο και να δει κανεί ποιες είναι οι επιπτώσεις της κατασκευής αυτών των φραγμάτων. Συμφωνώ και υπάρχει συζήτηση σε μικρό επίπεδο για την υδροελεκτρική ενέργεια, για εγκαταστάσεις υδροελεκτρικής ενέργειας και πώς μπορούν να υποστηριχθούν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, σχετικά το πώς ε, οι εγκαταστάσεις αυτές ε, θα μπορούσαν να βοηθήσουν μαζί σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις και επίσης και με τον ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας έχει δυνατότητες να έχει τέτοιες εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας. Ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες για αυτήν την μελέτη ε, σχετικά με τον προβληματισμό που υπάρχει για τις πολιτικές αυτές. Και τώρα φτάνουμε στο σημείο 6. Το θέμα είναι το άσυλο και μετανάστευση. Και η Μισελ ε, Στίφλερ ε, είναι η συγγήτρια. Άσυλο και μετανάστευση. ήταν θέματα καθαρά εσωτερικά ως προς την αντίληψή του. Σήμερα έχουν λάβει όμως και μία εξωτερική διάσταση στην δράση για της χρηματοδότησης Ένωσης. Κυρία Στρίφλερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, για τα θέματα τα σχετικά με, για τα εσωτερικά θέματα η Κομισιόν αποφάσισε να μειώσει τα προγράμματα στη διάρθρωση των δύο πυλώνων και για τη μετανάστευση και για την ε, εσωτερική ασφάλεια. Το Ταμείο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση θέλει να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις μεταναστευτικές ροές στην Ένωση, να ενισχύσει και να αναπτύξει το κοινό δίκτυο ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά η ολοκλήρωση και ενσωμάτωση των ε, πολιτών τρίτων χωρών στις χώρες της Ένωσης και μετά λογικές και αποτελεσματικές πολιτικές επιστροφής. Όλα αυτά για να μπορέσουμε να καλύψουμε, έχουμε ένα κονδύλι για να καλύψουμε τις δραστηριότητες ε, στις ε, τρίτες χώρες. Το Ταμείο επιτρέπει να χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεις στις τρίτες χώρες διασφαλίζοντας ε, τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τη συνέχεια ε, με τις ε, δράσεις που διαμείβονται στην επικράτεια της Ένωσης. Να συνδέσουμε δηλαδή καλύτερα την εσωτερική και εξωτερική διάσταση των εσωτερικών θεμάτων. Ας πούμε δράσεις οι οποίες ξεκινάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά πολύγουν στην τρίτη χώρα για την επιστροφή. Το θέμα της ε, κατάρτισης ε, των ε, νόμιμων μεταναστών προς την Ευρω... όταν μεταναστεύουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά είναι στα πλαίσια των αναπτυξιακών πολιτικών. Ο στόχος των ταμείων θα πρέπει να ε, αναπτύσσεται μέσα από τη συνένεση, την Ευρωπαϊκή Συνένεση για την ε, ανάπτυξη και τη συνεργασία. Και η ανάπτυξη και η συνεργασία θα λαμβάνεται υπόψη και ο εγκάρσια όλες τις πολιτικές για να καλύπτονται οι αναπτυσσόμενες χώρες. Έχω πολλές τροπολογίες που σε αυτή την κατεύθυνση στην εκθεσή μου. Οι άλλες αφορούν στην ανθρωπιστική βοήθεια. Το Ταμείο προβλέπει επιπλέον υποστήριξη για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε μέσα από κατεπίγουσα βοήθεια σε κατεπίγουσες ανάγκες ε, όταν τρίτες χώρες υπόκεινται έντονες μεταναστευτικές πιέσεις και οι δράσεις ε, που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία προς τις χώρες είναι συμπληρωματικέ με την υπόλοιπη πολιτική της Ένωσης και φυσικά και σέβονται την Ευρωπαϊκή κοινωνική για την ανθρωπιστική βοήθεια. Τώρα, για την οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, των διεθνών οργανώσεων, της ε, τοπικής κοινωνίας κλπ. Ε, αυτό θα μας επιτρέψει κατά τον προγραμματισμό να έχουμε αποτελεσματικότερη ε, αποτελεσματικότερα σχέδια και να έχουμε και μια πιο συμμετοχική διαδικασία. Πολλές χώρες ε, υποφέρουν ιδιαίτερα από την διαφυγή εγκεφάλων. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και να μπορέσουμε να το προβλέψουμε αυτό το στοιχείο και όταν αντιμετωπίζουμε την νόμιμη μετανάστευση. Ευχαριστώ ο κύριος Κόρτες Λάστρα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Στρίφλερ και για την πρόταση σχετικά με την μετανάστευση και το άσυλο που συμμερίζομαι. Ξέρετε όμως ότι η μετανάστευση και το άσυλο αποτελούν θερμόμετρο για την, την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Διότι νομίζω ότι στο δομέα της ανάπτυξης θα μπορούν, είναι, στα πλαίσια της ανάπτυξης έχουμε τον καλύτερο χώρο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό του είδους τα θέματα. Όταν εμείς ε, θέλουμε να ορίσουμε ένα ταμείο για τη μετανάστευση και το άσυλο, θα, μας, ε, θα πρέπει να έχουμε μία σοβαρή εστίαση για το τι σημαίνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να διέπει όλης αυτής, όλου αυτού του προγραμματισμού. και τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και, η και τα, Εθνικά Κοινοβούλια αλλά και οι άλλες, ε, τα κοινοβούλια των τρίτων χωρών και αυτά θα πρέπει αντίστοιχα να ρυθμίσουν. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει μία βελτίωση ως προς τις σχέσεις, αλλά να θυμίσω ότι η αναπτυξιακή βοήθεια δεν θα πρέπει με τίποτα να ε, συνδέεται με τη σύναψη συμφωνιών για την ε, διασυνοριακή συνεργασία, την απέλαση ή την υποδοχή. και θα πρέπει να απαιτήσουμε να υπάρξει μια πολιτική διεθνών προδιαγραφών για το θέμα της υποδοχής των μεταναστών στις τρίτες χώρες. Κυρία Σνίμπερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τη συνάδελφό μου. Είναι πάρα πολύ καλή η έκθεση. Θα ήθελα ρητά να την ευχαριστήσω για τις καλές ε, προτάσεις της. Καταρχάς, για την συνοχή της πολιτικής γενικότερα, αλλά και για τη τόσο σημαντική συνέργεια μεταξύ των διαφόρων ταμείων που μας περιέγραψε και τόνισε ιδιαίτερα η Μισελ Στρίφλερ. Ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Ο Κάρλος Καρδάου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχά, ε, Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις τροπολογίες που κάνετε και τις προτάσεις σας. Κυρία Συγκητρία. Στην παρούσα φάση μπορούμε να πούμε ότι ορισμένες ε, ε, είναι πάρα πολύ ευπρόσδεκτες και μάλιστα βελτιώσουν και τη διατύπωση για τη συνέχεια και συνεκτικότητα της πολιτικής για την αναπτυξιακή ανθρωπιστική βοήθεια. Μπορούμε να εξετάσουμε τις δυνατότητες που έχουμε, να προσαρμόσουμε τη διατύπωση των αιτιολογικών σκέψεων για να ενισχυθεί αυτή η συνέργεια και η σημασία για να υπάρχει και μια συνοχή μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής και προκειμένου με την ε, απτυξιακή βοήθεια. Έχουμε περισσότερες αιτιολογικές σκέψεις που αναφέρονται σε αυτή. Βεβαίω θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τη διατύπωση. Γίνονται κάποιες προτάσεις χωρίς να προεξοφλώ και με την επιφύλαξη των όσων θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν θα πρέπει σε όλα τα άρθρα, όπως προτείνετε στην έκθεσή σας, να επαναλαμβάνουμε ε, την συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής δεν είμαι βέβαιος δηλαδή αν θα πρέπει στο διατακτικό σε κάθε άρθρο να τα λέμε αυτά. Δεν φτάνει να το κάνουμε μόνο στις αιτιολογικές σκέψεις. Θα το επανεξετάσουμε, όμως θα προβούμε σε αναδιατυπώσεις και θα επανέλθουμε στο κοινοβούλιο. Επίσης, τίθεται το θέμα της διαβούλευσης και της εταιρική σχέσης και προτάθηκε. Μάλλον αναφέρθηκε η δυνατότητα διαβούλευση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από τη φάση του σχεδιασμού μέχρι την αξιολόγηση, την εκτίμηση και τον έλεγχο και την παρακολούθηση ε, κοιό και αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης της Ένωσης αλλά και τρίτων χωρών. Βεβαίως μπορούμε να μελετήσουμε αυτό το ενδεχόμενο, αλλά είναι μάλλον θέμα έτσι εγκάρσιο. Έχουμε τέτοιες ε, συστάσεις για άλλα μέσα και αυτό που θα ήθελα να σας πω εδώ είναι ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όντως θέλουμε να έχουμε αυτή τη δυνατότητα χρηματοδότησης κάποιων δράσεων εκτός της Ένωσης, αλλά θα είναι πάρα πολύ περιορισμένες στο πεδίο εφαρμογής τους και όπως εξηγεί η εισηγήτρια για την εξυπηρέτηση κυρίως κοινοτικών συμφερόντων. Ε, για κάποια θέματα που έχουν άμεση επίπτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν σε ποιο βαθμό δικαιολογείται να γίνει διαβούλευση εταιρική σχέση με οργανώσεις τρίτων χωρών. Γιατί υπάρχουν και πρακτικά ζητήματα εδώ. Και σε ποιο βαθμό δηλαδή μια τέτοια διαβούλευση δικαιολογείται στα πλαίσια του παρόντος μέσου. Εγώ δεν είμαι καν σε θέση να σας δώσω την άποψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά. Απλώς σημειώνουμε τις προτάσεις σας και επιφύλασσόμεθα. Επίσης η διαφυγή εγκεφάλου είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για μας και μας απασχολεί. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε και από πλευράς διατύπωσης να το ρυθμίσουμε. αλλά και πάλι όχι στο διατακτικό, ε, ενδεχομένω στις αιτιολογικές σκέψεις, εκεί που αναφέρουμε τις γενικές αρχές εφαρμογής αυτών των μέσων, αυτού του μέσου. Και όταν μιλούμε για την νόμιμη μετανάστευση και πώς μπορεί αυτή να υποστηριχθεί, θα μπορούσαμε να σημειώσουμε και εκεί τη σημασία του θέματος της διαφυγής εγκεφάλων. Σταματώ εδώ, αν έχετε ερωτήσεις είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Στρίχλερ για να απαντήσει. Να σας πω ότι κατανοώ τις ανησυχίες σας. Να δούμε τι θα μας πει η Κομισιόν. Αλλά εγώ είμαι... Εγώ προτιμώ να επαναλαμβάνουμε τα πράγματα για να είμαστε σίγουροι δηλαδή ότι τα έχουμε μέσα. Δηλαδή Δεν ξέρω, το να μη λέμε μερικά πράγματα μόνο και μόνο για ευχαρίστηση, δεν ξέρω, ας περιμένουμε την Κομισιόν. Εγώ προτιμώ να λέω τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Περνάμε ίσως στο θέμα το οποίο είναι το πιο σημαντικό για τη σημερινή μας συνεδρίαση. Στην έκθεση του κυρίου Τίσμπερμαν για την ε, δημιουργία χρηματοδοτικού μέσου για την αναπτυξιακή συνεργασία. Πολλοί μήνες ε, ε, πυρετόδους εργασίας σχετικά στην ομάδα εργασίας και ο εισηγητής μας, ο κύριος Μπέρμαν, θα μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσης που έχει τις τελευταίες προτάσεις του, όχι μόνο για τις επόμενες πολιτικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής συνεργασίας, αλλά και για αποτελεσματικές διαδικασίες και μια πραγματική εμπλοκή κοινοβουλευτική συμμετοχή κοινοβουλευτική στην λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Θα έχουμε και γνωμοδότηση τεσσάρων άλλων επιτροπών των οποίων ε, οι εισηγητές οι αντίστοιχοι κλήθηκαν να λάβουν μέρος σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Δίνω λοιπόν το λόγο στον εισηγητή για να μας παρουσιάσει αυτή την έκθεση. Κύριε Μπέρμαν, σας δίνω το λόγο. Ναι, κυρία Πρόεδρε, πόσα λεπτά έχω για αυτήν την παρουσίαση. Ε, όλο το χρόνο που θέλετε. Δεν υπάρχει σημαντικότερο θέμα στη θητεία μας από το θέμα αυτό. Έχουμε προβλέψει μία ώρα για σας, κύριε Μπέρμαν. Πολύ καλά. Λοιπόν, προσοχή. Στα αγγλικά λυπούμε. Ε, το μέσο αναπτυξιακής ε, συνεργασίας ε, είναι στο επίκεντρο του προϋπολογισμού για να συμμετάσχουμε στην παγκόσμια τάξη και στο ίσο δικαίωμα κάθε πολίτη του κόσμου για κράτος, δικαίου, δημοκρατία, καλή διακυβέρνηση και η φόρο ανάπτυξη. Με αυτές τις υψηλές φιλοδοξίες διάβασα ε, για το 2014-2020 την πρόταση ε, της ε, Κομισιό για το μέσο αυτό αναπτυξιακής συνεργασίας. Πιο απλό, πιο σαφές και κάνει διάκριση ανάμεσα στις τοχότερες χώρες και στις χώρες που γίνονται αναδυόμενες οικονομίες. Ένα νέο βήμα στον προγραμματισμό των κρατών μελών και της Κομισιό. Η ευθυγράμμιση, η οικειοποίηση είναι, αρχέ αρχές οι οποίες υιοθετήθηκαν και επίσης η αρχή της καλύτερης εστίασης η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συγκεντρωθεί σε τρεις τομείς στο μέγιστο αναχώρα. Επίσης προσφέρει νέες, ε, νέες ε, ε, διαδικασίες ανάμειξης. Υπάρχει λοιπόν σε, αυτήν, αυτό το μέσο, τη ΜΑΣ, στο Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας, νέες προτάσεις χάρη στην, στην ομάδα αυτή που είναι διοικητική μπόρεσα να καταθέσω πάνω από 200 τροπολογίες. Μην γελάτε, μην γελάτε είναι σοβαρή εργασία, σοβαρή. Οι τροπολογίες αναφέρονται κυρίως στην εφαρμογή των αρχών ε, του ΜΑΣΑ ε, και νέες προσεγγίσεις, πιο προσεκτικές, ε, πιο ριζικές. Οι τροπολογίες έχουν πολλούς στόχους. Πρώτον, η κατουξιοδότηση πράξης με τους εισηγητές και άλλα μέσα. Ο εισηγητής εισάγει το μέσο των κατουξιοδότηση πράξεων για την ταχύτητα των αποφάσεων όπως επίσης και την, ε, το δημοκρατικό έλεγχο από αυτό το κοινοβούλιο. Σαφήνια για τις δράσεις που προβλέπει αυτό το μέσο. Αυτός ο μηχανισμός, βεβαίως ενώ η Κομισιόν χρειάζεται μια ευελιξία, ε, η διατύπωση χρειάζεται κάποια αναθεώρηση, όπως λέξεις όπως where, as και inter στα αγγλικά έχουν διαγραφεί. Αλλιώ θα ήταν ένα, μια επιταγή εν λευκό για την Επιτροπή με τις ε, τροπολογίες ε, μπορούν ε, ε, έχουμε μια σχέση ανάμεσα στην αρρωγή, στην αποκατάσταση και στην ανάπτυξη. Επίσης η κατεπίγουσα διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με έγγραφα προγραμματισμού. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία αυτή δεν, ε, δεν εμποδίζει την ε, Κομισιόν να λάβει κατεπήγοντα μέτρα. Επίσης, στο παράρτημα διευκρινίζονται τα, οι δράσει στα γεωγραφικά προγράμματα. Βάσει τη τροπολογία μα, στο Ευρωπαϊκό Κονσένσου για την Ανάπτυξη και έλαβα υπόψη τον κανονισμό για το ΜΑΣ που έχουμε, όπως και τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι θέσεις για τις διάφορες περιφέρειες. Η διαφοροποίηση ανάμεσα στους πτωχούς και τους λιγότερο πτωχούς. Δεν έχει κανένα νόημα ε, να συνεχίζουμε προγράμματα με χώρες που μπορούν να αγοράσουν βαλιστικούς πυράβλους και σοβαρούς εξοπλισμούς. Συμφωνούμε ότι οι πτωχότερες χώρες θα πρέπει να δικαιούνται υψηλότερα κονδύλια. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των αναπτυσσομένων χωρών για τα γεωγραφικά προγράμματα είναι το ΑΕΠ ανακεφαλή. Αλλά πιστεύω ότι η κοινωνική ανισότητα θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη και προσίζω, ε, προτείνω τέσσερα πρόσθετα κριτήρια. Ο δείκτης ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού, το κεφαλή δείκτης φτώχειας, ο δείκτης χάσματος φτώχειας ε, και επίσης ο συντελεστής ε, τζίνι του εισοδήματος. Εκτός αυτού και εύχομαι τύχη στους μεταφραστές για να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα ή τα προγράμματα αναχώρα θα πρέπει να συγκεντρώνουν σε χώρα όπου έχει μοχλό πίεση η τα προγραμματα αναχωρα θα πρεπει να συγκεντρωνε σε Ένωση και προσφέρει ε, προστιθέμενη αξία για την μείωση της φτώχειας και του χάσματος. Ο κατάλογος μας είναι μακρύτερος των μέτρων από τις Κομισιόν για χώρες που δεν είναι επιλέξιμες για διμερή συνεργασία. Ε, προτείνω ε, προοδευτικά να υπάρχει μια διαδικασία. Μια τέτοια εξάλληψη προοδευτική είναι μια επιλογή και μια εξαίρεση και δεν πρέπει να ισχύει για όλες τις χώρες. Βεβαίως είμαι ανοιχτό σε προτάσεις και βελτιώσεις ε, και μπορούμε, πρέπει όμως να συγκεντρωθούμε σε κριτήρια και στόχους και όχι σε μεμονωμένες χώρες ο εισηγητής εισήγαγε διάφορες τροπολογίες που ενισχύουν ε, την προσέγγιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε αυτήν την πολιτική προοπτική η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποδείξει την προστιθέμενη αξία, να μην είναι ο ως όγδος ε, δωρητής, ε, αλλά να, ε, να έχει την υποστήριξη των κρατών μελών. Έχουμε την αλλαγή από την Κομισιόν για την αρχή ότι τουλάχιστον 20% του προϋπολογισμού του κανονισμού αυτού να χρησιμοποιείται για εκπαίδευση και υγεία, όπως είναι με το μέσο που έχουμε τώρα. Πρόταση της Κομισιόν είναι να διευρυνθεί και να γίνει 20% για ανθρώπινη ανάπτυξη και δεν έχει κανένα επιχείρημα γι' αυτό και αυτό καλύπτει ευρύ φάσμα δράσης από την ε, εκπαίδευση ως το οικονομική ανάπτυξη. Θέλουμε να μειώσουμε αυτό το φάσμα, να έχουμε 20% για κοινωνικές υπηρεσίες σύμφωνα με τους ορισμούς των Ηνωμένων Εθνών στους στόχους της χιλιατίας, στους αναπτυξιακούς σχετικά με το Παναφρικανικό πρόγραμμα ενός δισεκατομμυρίου προσπάθησα να διευκρινίσω τους τομείς δράσης που πρέπει να καλύπτει το πρόγραμμα μέσα στο κονσένσους για την ανάπτυξη. Ελπίζω ότι η ε, συζήτηση αύριο θα επιτρέψει μεγάλη συνεισφορά και συμβολή για νέες τροπολογίες. Μια άλλη πτυχή είναι η σχέση ανάμεσα ε, στην σύνδεση αρρωγής αποκατάστασης και ανάπτυξης για ανθρωπιστικούς τομείς. Θα πρέπει το χάσμα να μειώσει και η σύνδεση να είναι μεγαλύτερη, να ενισχυθεί ο ρόλος ε, των οργανώσεων ε, της κοινωνίας των πολιτών. Επίσης τονίζω την σημασία των ευάλωτων και παραμελημένων ομάδων όπως είναι οι γυναίκες, τα παιδιά, τα κορίτσια, τα άτομα με αναπηρίες, οι μειονότητες και ε, το τμήμα ε, πολιτισμού επίσης έχει προσθεθεί ο εισηγητής ήδη συζήτησε εντατικά με την Κομισιόν και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και περιμένει συνέχιση αυτής της συνεργασίας ώστε να αποφευχθούν πολλές γκάφες και λάθη. Ε, και αφήνω τα θέματα αυτά στην Κομισιόν. Προς τους κοιόδη εισηγητές ε, ήμουν σε στενή επαφή με όλους από την αρχή της εργασίας αυτής και θα εξακολουθήσω τη συνεργασία μέσα στο ίδιο πνεύμα. Ευχαριστώ. Thank you. for this very... Ευχαριστώ για αυτήν ε, την εντατική εργασία και τις 200 τροπολογίες. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό. αυτά, ο κύριος Γκόρενς έχει τον λόγο. Προτού... Προτού αντιδράσω, ευχαριστώ τον Τάις Μπίρμαν για την, για την παρουσίασή του, που μπόρεσα εν μέρη να παρακολουθήσω. Τώρα μίλησες για τη διαφοροποίηση. Τι αλλάζει. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των προτάσεών σου και των προτάσεων της Κομισιόν. Όταν παίρνουμε μόνο το ΑΕΠ μιας χώρας, βλέπουμε μόνο το μισό του ΑΕΠ επί του πληθυσμού. Δεν βλέπουμε τις κοινωνικές ανισότητες. Διότι πολλές φορές ο πλούτος μιας χώρας μπορεί κάλλιστα να συγκεντρώνεται στο 5% του πληθυσμού. Και γι' αυτό προτείνω να προσθέσουμε αυτά τα τέσσερα κριτήρια. Η Κομισιόν. Δεν ξέρω ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Ε, Λουκ Μπαγκίο από την Η Κομισιόν εφράζει την ικανοποίησή της για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί του θέματος και εδώ και στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο στις 25 Ιουνίου ενέκρινε τη γενική προσέγγιση της Κομισιόν και ελπίζουμε στις αρχές Οκτωβρίου να ξεκινήσουμε τον άτυπο τρίλογο. Έχουμε, συγκλίνουμε σε πολλά σημεία και σε πολλά σημεία υπάρχει και συνένεση. Ας πούμε για τον κοινό προγραμματισμό μεταξύ κομισιών και κρατών μελών, επιγράμμιση των πολιτικών, ε, των κρατών, ε, εταίρων κλπ. Αυτή είναι η ενίσχυση επίσης ε, των αναφορών για, για τον σεβασμό των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος, δικαίου, δημοκρατία κλπ. Τώρα για τις διαπραγματεύσεις του μέλλοντος να σας εκφράσω και εγώ μερικές ανησυχίες της Κομισιόν. Πρώτο, έχουμε την αρχή διαφοροποίησης είναι ένα από τα σημεία κλειδί της ε, έκθεσής της. Εμείς θεωρούμε ότι 11 χώρες που έχουν ένα εισόδημα 19 ε, χώρες ε, οι οποίες βρίσκονται σε μία μέση κατάσταση μπορούν κάλλιστα να τα καταφέρουν χωρίς να παίρνουν αναπτυξιακή βοήθεια για να καταπολεμήσουν τη φτώχεια. Τώρα η θέση της Κομισιόν ήταν να είναι δεσμευμένη πάντοτε με τις ε, χώρες εταίρους, ε, δεσμευμένη και σε περιφερειακά προγράμματα για ειδικέ προβληματικές ε, των ενδιαφερομένων περιφερειών, όπως επίσης και θεματικά προγράμματα υποστήριξη για τη δημοκρατία, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την κοινωνία των πολιτών για την ε, καταπολέμηση της τροφιμικής ασφάλειας. Υπάρχει λοιπόν μια σχετική συνένεση μεταξύ των οργάνων για να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαφοροποίηση. Αλλά εμείς ε, θεωρούμε με τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου ότι η αρχή της διαφοροποίησης κάπως διαχέεται, αποδυναμώνεται. Για παράδειγμα, εμείς ας πούμε για το θέμα των ε, διαφόρων ε, συνεργασιών και των όρων σύναψης συνεργασίας, θεωρούμε ότι με, με, με τις τροπολογίες που προτείνεται θα μπορούσαμε κάλλιστα να, αν τις ερμηνεύσουμε με έναν τρόπο, να επιλέξουμε και τη Βραζιλία. Ε, η ενίσχυση τώρα, της, η αύξηση ενίσχυσης ανατοχ, χρονικά ε, χωρίς να υπάρχει η αρχή της ερετιμότητας, χωρίς να έχουμε τελειοποιημένο phasing out, ε, δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι αυτές οι χώρες ε, μπορεί ναι, να, να είναι φτωχές, αλλά δεν θα πρέπει να εξαρτώνται 100% από την εξωτερική βοήθεια. Θεωρούμε ότι μπορούμε να βρούμε λύσεις για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανοσοχίες της της Επιτροπής σας, κυρίως για τις χώρες των άνδεων. Ένα δεύτερο σημείο ανησυχίας είναι στο πολιετές πλαίσιο. Εδώ δεν θα σταθώ γιατί πρόκειται για ένα οριζόντιο επίπεδο, αφορά και άλλα ε, θέματα που αφορούν και στον τίτλο 4 αλλά και τις εσωτερικές πολιτικές. Μιλάω εγώ για τις ενταλμένες πράξεις τα θέματα στρατηγικής έτσι όπως προβλέπονται από την πρόταση της Κομισιόν για τη μορφή τους και για το περιεχόμενό τους δεν εντάσσονται μέσα από αυτή τη διαδικασία των δεταλμένων πράξεων και η διαδικασία της επιτροπολογίας είναι αυτή που πρέπει να εφαρμόζεται. Θα επανέλθουμε όμως αυτό για το, κατά το μέλλον των διαπραγματεύσεων διότι είναι ένα θέμα κεντρικό. Ένα τελευταίο σημείο ανησυχίας αφορά στη συγκέντρωση της βοήθειας. Εμείς ε, θεωρούμε θεωρούμε ότι πάντα θα πρέπει να έχουμε προτεραιότητα για την ανάπτυξη θεωρούμε ότι ένας κατάλογος αναλυτικός ε, θα ήταν καλύτερος για την ενίσχυση της αναπτυξιακής πολιτικής. Άλλα σημεία που θεωρώ ότι είναι προβληματικά και πρέπει να συζητήσουμε στο μέλλον είναι η μείωση της ευελιξίας για το Παναφρικανικό προγράμμα. Εμείς είχαμε προτείνει 10% ευελιξία, είχαμε προτείνει 10, λοιπόν μας το μειώσανε στο 5% για το Erasmus for All είχαμε ένα 2% ως ποσό αναφοράς το οποίο όμως φαίνεται να είναι και μικρότερο, αλλά λάβουμε υπόψη της δράσης στο παρελθόν. Ο κύριος Γκέρετς πάλι. Ε, διαπιστώνω ότι έχουμε πρόβλημα στη διαφοροποίηση. Ο ΤΕΙΣ έχει δίκιο στην ανάλυση του όταν διαπιστώνει ότι εκείνοι που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη ε, ε, ενίσχυση ε, από το κράτος και από τις αναπτυξιακές βοήθειες είναι εκείνοι που πλήττονται από τις ανισότητες. Μα αυτό είναι πολιτική επιλογή. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε την δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια σε συνάρτηση των ανισοτήτων, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως πριμοδότηση της ανευθυνότητας ε, των δικαιούχων ε, χωρών. Δηλαδή, όσο λιγότερες προσπάθειες έκαναν για την αναδιανομή του πλούτου, τόσο περισσότερο ε, υπό τη δική του αντίληψη δικαιούνται δημόσια βοήθεια. Και εδώ εξηγείται η αρχή της διαφοροποίησης στην προτείνει Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος να ξεφύγουμε από αυτό είναι να ε, ε, κινήσουμε μια πραγματική πολιτική συζήτηση και ε, να φέρουμε ενώπιον των ευθυνών τους τα κράτη που ευθύνονται για αυτές τις ανισότητες και να μας εξηγήσουν λίγο τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να ξεπεράσουν αυτές τις δυσκολίες. Εκεί έχουμε πρόβλημα και η διάσκεψη του ερχομένου Σεπτεμβρίου για τους στόχους της χιλιετίας για την ανάπτυξη, ε, περί αυτού θα ε, στραφεί. Θα πρέπει όλοι να έρθουν ενώπιον των ευθυνών τους και οι αναδυόμενες χώρες. Λέει, ακόμα και αν ξεπεράσουμε το 0,7% δεν πρόκειται να ξεφύγουμε αν δεν κάνουν τίποτα οι χώρες ενός μέσου εισοδήματο. Συμφωνώ με 90% των όσων προτείνει ο ΤΑΙΣ στην εξαιρετική του κατά τα άλλα έκθεση, αλλά σε αυτό το θέμα της διαφοροποίησης θα πρέπει να ξανανοίξουμε τη συζήτηση, γιατί απέχουμε έτη φωτός από την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και όλοι με πολύ εύσχυμο τρόπο προσπαθεί ε, προσπαθούν να προφασιστούν μια συνένεση ανύπαρκτη. Κύριε Μπέρμαν, έχετε το λόγο αν θέλετε για να απαντήσετε και να κλείσετε. Κοιτάξτε, αυτά είναι ακόμα στο στάδιο της εκπόνησης. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας, είναι πάρα πολύ ε, Για το θέμα της συνένεσης που προφασίζεται ή δείχνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχετε δίκιο. Υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία συμφωνούν το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο ε, ως προς την προσέγγιση της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για το θέμα ότι μας δικάζουν διάφορα θέματα, επίσης έχετε δίκιο, για, για τις κατεξουδότηση πράξεις θα έχουμε ε, συζήτηση εκτενέστερη. Το είπε και ο Σαλ Γκέρενς, θα πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθούμε με τις ανισότητες, αλλά δεν πιστεύω ότι κάτι τέτοιο σημαίνει επιβράβευση ή πρημοδότηση ε, της έλλειψης ε, καλής διακυβέρνησης. Νομίζω αυτό είναι λίγο τραβηγμένο. Θα πρέπει όμως να συνεχίσουμε τη συζήτηση για τη διαφοροποίηση και θα βρούμε έναν τρόπο να βγούμε από αυτή τη σύγκρουση για το θέμα. Γιατί επί της αρχής συμφωνούμε όλοι. Και επίσης συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πολλές χώρες θα μπορούσαν να αφαιρεθούν από τον κατάλογο και να είναι επιλέξιμες για διμερή βοήθεια Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει συνένεση επί της αρχής. Δεν νομίζω ότι τα νέα κριτήρια είναι ε, υπερβολικά περίπλοκα. Είναι πιο εξειδικευμένα από το απλό κριτήριο του Ε.Π. Θα δω τις τροπολογίες των συναδέλφων ε, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και μετά θα αρχίσουμε τη συζήτηση για την τελική διατύπωση της έκθεσης με τις τροπολογίες των συναδελφών. Αυτό είναι πολύτιμο, επαναλαμβάνω. Θα συνεχίσουμε ε, τι επαφέ και τι συζητήσει με το Συμβούλιο, την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να είναι η έκθεση καλύτερη, δυνατή τελικά. Ευχαριστώ πολύ. Deja pasar este momento para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 Η Κομισιόν ζητά μία ευελιξία. Να μπορούμε δηλαδή να ξοδεύουμε κονδύλια τα οποία δεν αποτελούν τμήμα κατά 10% που δεν αποτελούν τμήμα της επίσημης ε, αναπτυξιακής βοήθειας αντί του 5% που προτείνω εδώ. Εμείς ε, θέλουμε να προστατεύσουμε την Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Βοήθεια, η οποία δέχεται μονίμως επιθέσεις με αυτή την τροπολογία. Θέλουμε, λοιπόν, θεωρούμε, θεωρώ ότι αν αφήσουμε την ευελιξία κατά 10%, ε, θεωρητικά, η Κομισιόν ποτέ δεν θα το καλύψει αυτό το ποσοστό, διότι το ποσοστό είναι πολύ χαμηλότερο και το 5% δεν φτάνει δηλαδή, άρα κάλλιστα μπορεί να επιβιώσει η Κομισιόν με το 5%. Για, το, ε, ε, για τον έρασμο, 10%, το 2% του προϋπολογισμού μας για αυτό το σκέλος του προγράμματος θα μειώσει συνολικά τον προϋπολογισμό του έρασμου. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε μία συνεδρίαση με όλους τους συνεισηγητές για την χρηματοδότηση και να συμφωνήσουμε για ένα ποσοστό προς στιγμήν. διότι το δικό μας ταμείο, το DCI, συμμετέχει κάπως δυσανάλογα σε όλη αυτή την ιστορία. Γι' αυτό βάλαμε εμείς αυτό το ποσοστό 2%. Εγώ είμαι έτοιμος να το συζητήσω με όλους τους συνεισηγητές για τα χρηματοδοτικά μέσα από τις άλλες επιτροπές. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκέρεντς, δεν σας είχα δει. Σχετικά με τον έρασμο, εγώ θεωρώ ότι όλο το τμήμα προπολογισμού το οποίο ε, χρεώνουμε στο DCI για τον έρασμο όπου DCI χρηματοδοτικό μέσο για την ανάπτυξη, DCI προσυντομία. Δηλαδή, όλα τα κονδύλια τα οποία θα παίρνουμε από το DCI θα πρέπει να είναι πάντοτε κονδύλια για την ανάπτυξη. Δηλαδή να πούμε ότι δεν θα αποδυναμώνουμε την ανάπτυξη αφαιρώντας τις κονδύλια. Λοιπόν, πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα λέει η Πρόεδρος, θα το συζητήσουμε και αύριο. Λοιπόν, διακόπτουμε τώρα τη συνεδρίαση. Θα συνεχίσουμε αύριο στις 10. Τώρα θα συνεδριάσουν οι συντονιστές και κλεισμένων των θυρών. Αύριο θα αρχίσουμε με μία ψηφοφορία. Σας θυμίζω ότι θα πρέπει να φέρετε τις μαγνητικές σας κάρτες.